Uh, good uh, gentlemen. Uh, let me welcome. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς, σας καλωσορίζω στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας και καλωσορίζω και δύο προσώπους της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας, την κυρία Τεμενούζκα Πέτκοβα και τον κύριο Ιβάιλο Μοσκόφσκι. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχουμε τον πρώτο μήνα της ε, Βουλγαρικής ε, Προεδρίας, Συγχαρητήρια και κοιτάω και την γραβάτα σας κύριε Υπουργέ. Α, δεν είναι η επίσημη γραβάτα. Οι Βούλγαροι όμως ε, συνάδελφοι και εγώ έχουμε την επίσημη γραβάτα της Προεδρίας. Ε, συμβολικό νομίζω. Και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτά τα σύμβολα. Είναι νομίζω ένα μικρό σημάδι, αλλά πολύ σημαντικό. Και πολύ ωραία γραβάτα κιόλα. Και σα συγχαίρω για το γούστο σα. Περνάμε τώρα στην ακρόασή μας. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι πολύ απλή. Πρώτα απ' όλα, να ζητήσω από εσά τους δύο υπουργούς, την κυρία Πέτκοβα, την Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών και Πυρηνικών Ζητημάτων επίση και τον κύριο Μοσκόφσκι, τον Υπουργό Μεταφορών, Τεχνολογίες, Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω τον λόγο για 7 λεπτά λίγο πολύ και μετά να γίνει μια συζήτηση με τους βουλευτές και στο τέλος ε, της συζήτησης αυτής ε, θα θέλαμε τις δικές σας απαντήσεις. Στις 6.30 λίγο πολύ. Στις 4.30 με συγχωρείτε θα συναντήσουμε τους δύο επόμενους υπουργούς οικονομίας ε, και παιδείας. Τέσσερις συνολικά υπουργοί σήμερα το απόγευμα. Αυτά λοιπόν νομίζω ως εισαγωγή. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις αρμοδιότητές μας εδώ. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα κάνατε. Κυρία Πέτκοβα. Και αναμένουμε να ακούσουμε τις προτεραιότητές σας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούζεκ, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη τιμή και ευχαριστήση για μένα να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλευτικής Προεδρίας του Συμβουλίου στον τομέα της ενέργειας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ιδιότητά του συνομοθέτη. Πριν από σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας να ασκήσουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τεράστια ευθύνη και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι συνειδητοποιούμε την ευθύνη αυτή. Το κύριο καθήκον μας θα είναι να αναζητήσουμε συμβιβασμούς και ομοφωνία προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Για μας ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υψίστης σημασίας. Γνωρίζουμε ότι μόνο με επικοδομητικό διάλογο μπορούμε να επιτύχουμε τους κυρίους στόχους και τις προτεραιότητές μας. Ως Προεδρία αντιμετωπίζουμε πολλές και διάφορες προκλήσεις. Αυτό κυρίως ισχύει για τον ενεργειακό τομέα. Και είναι και κατανοητό. Γιατί αυτός ο τομέας είναι πολύ σημαντικός ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Ανάλογα με το πώς αναπτύσσεται το τομέας, ε, μπορεί να δούμε ευημερία στις οικονομίες μας ή μπορεί και όχι. Κατόπιν της ε, τεράστιας επιτυχίας της Εσθονίας, Και εμείς ανυπομονούμε να εργαστούμε εντατικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πλειονότητα των φακέλων που αφορούν το πακέτο της καθαρής ενέργειας για όλους τους Ευρωπαίους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η βουλγαρική κυβέρνηση και η βουλγαρική προεδρία είναι έτοιμες για επικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βάλουμε τα δυνατά μας ε, προκειμένου να καταλήξουμε στους απαραίτητους συμβιβασμούς από κοινού. Ο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε τις κυρίες προτεραιότητές μας στις ε, διαπραγματεύσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσουμε τις ε, αρχές της Ενεργειακής Ένωσης. Ε, θέλουμε να έχουμε ενέργεια φτηνή και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους Ευρωπαίους. Η Ενεργειακή Ένωση μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο αν λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Είμαι σίγουρη κυρίες και κύριοι πως αυτή η δεσμή μέτρων για την ενέργεια είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και μοναδική. Γι' αυτό συνειδητοποιούμε ότι η επίτευξη συνένεσης μεταξύ των μελών και κοινοβουλίου δεν θα είναι κάτι εύκολο. Είναι μεγάλη πρόκληση που έχουμε ενωπιών μας, αλλά είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση μας και σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητές μας, θα ήθελα να αναφέρω τον ε, κανονισμό για τη χρήση της ενέργειας, την ε, οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, και έναν ακόμη φάκελο. Θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά άλλους νομοθετικούς φακέλους, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται χρόνο προκειμένου να καταλήξει σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς και θα χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για το αέριο, γνωρίζουμε ότι αυτός ο φάκελος είναι πάρα πολύ σημαντικός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα φάκελο που έχει μεγάλο αντίκτυπο σε όλα τα κρατη τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά αυτό το φάκελο. Ο κύριος μας στόχος θα είναι να πετύχουμε την συνένεση και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό τόπο μεταξύ των κρατών μελών. Τελικά, επιθυμούμε να έχουμε μια κοινή θέση στο φάκελο αυτό. Ποιες είναι οι κυρίες προτεραιότητές μας. Η κυρία μας προτεραιότητα είναι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων. Για μας είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε για την ε, διαφοροποίηση πηγών και οδών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Μιλώντας για ενέργεια και μιλώντας για τα κύρια στοιχεία του προγράμματος της Βουλγαρικής Προεδρίας θα ήθελα να αναφέρω την, ε, οικοδόμηση, την δημιουργία των ε, υποδομών που λείπουν σε αυτήν την περιοχή γιατί μόνο αν ε, φτιάξουμε αυτές τις υποδομές θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε τον ενεργειακό εφοδιασμό την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα για όλη την περιφέρεια. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, Γνωρίζω ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να σας παρουσιάσω τις κύριες μας προτεραιότητες. Ωστόσο, ανέφερα τα highlight της Βουλγαρικής Προεδρίας. Θα ήθελα βέβαια να δράξω την ευκαιρία για να τονίσω ότι θα είμαστε ένας αξιόπιστος εταίρος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος στόχος μας θα είναι να εργαστούμε προς ε, μια πιο ασφαλή και νοτόμο Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ιβάιλο Μοσκόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη μου τιμή να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη συνένεση, την ανταγωνιστικότητα και την συνέπεια για όλους τους τομείς. Ούτως ώστε να αναβαθμίσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια και έχουμε τις τέσσερις βασικές μας προτεραιότητες, τέσσερις άξονες γύρω από τους οποίους θα περισταθεί το έργο μας τους επόμενους μήνες το μέλλον της Ευρώπης, σταθερότητα, ασφάλεια, ψηφιακή οικονομία, ψηφιακές δεξιότητες καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική αλλά και την συνδεσιμότητα για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ένας από τους στόχους μας είναι μέχρι τέλος του έτους να έχουμε ολοκληρώσει την ψηφιακή αγορά. Και θα συνεχίσουμε το έργο μας με την ψηφιακή οικονομία, τις ψηφιακές δεξιότητες, ούτως ώστε να συμπληρώσουμε τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά. Και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας ούτως ώστε να υπάρχει ε, ε, κάποιο είδου συνέχεια μέσω της Τρόικα και να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα. Οπότε έτσι θέλουμε να επιταχύνουμε την ε, ψηφιακή τεχνολογία και να φτάσουμε στις τεχνολογίες πέμπτης γενεάς 5G και να υπάρχει και η πολυτροπική πρόσβαση. Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια συγκυρία κατά την οποία το θεματολόγιο είναι πολύ απαιτητικό σε σχέση με τα τρέχοντα εκκρεμούντα θέματα, σε σχέση με τις προσδοκόμενες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρόκειται να προβληθούν την Άνοιξη. Οπότε και φέτος την Άνοιξη αυτό το οποίο θα κάνουμε εμείς είναι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις που αφορούν την μεταρρύθμιση του κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου των επικοινωνιών. Αυτό που λέγεται κώδικας. Να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά και να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω που είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό θα καθορίσει τις εξελίξεις στον τομέα του ανταγωνισμού, τις επενδύσεις στο 5G και επίσης σε δίκτυα υψηλών δυνατοτήτων. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, οπότε και στο δικό μας θεματολόγιο έχει υψηλή προτεραιότητα. Θέλουμε επομένω μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά το σχετικό νομοθέτημα και έτσι η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΕΝΙΣΑ να μπορέσει να έχει μια διαρκή μόνιμη εντολή, μια στεγανή εντολή ούτω ώστε να μπορεί να δημιουργήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή επιστοποίηση. Αυτό θα εξασφαλίσει αξιοπιστία και ασφάλεια στο διαδίκτυο και πρόκειται επίσης να αντιμετωπίσουν την κατάτμιση της αγοράς που ισχύει σήμερα. Θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των μη προσωπικών δεδομένων που είναι πολύ βασικό για την ε, οικονομία των δεδομένων. Είναι και προϋπόθεση για την λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας και έτσι θα δημιουργούν θέσεις εργασίας. Έτσι θα καθοριστούν και ποιε θα είναι οι δείξοντε του μέλλοντος. Οπότε και έτσι με τα δεδομένα θα υπάρχει μια ελεύθερη διακίνησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ε, στην Ένωση σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και επίσης γνωρίζουμε ότι ο κόσμος χρειάζεται εμπιστευτικότητα, διαβάθμιση στα ηλεκτρονικά δεδομένα, χρειάζεται ηλεκτρονική και η προστασία του ιδιωτικού βίου, άρα θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της υπαρκούς προστασίας αλλά και της πρόθεσης της καινοτομίας. Κατά την Προεδρία μας ελπίζουμε να συζητηθεί η τρίτη δεσμεύον για τα δεδομένα τώρα το ότι θα πρέπει να ξανοιχθεί και ο δημόσιος τομέας. Ε, αυτό είναι κάτι αναμφίβολο όσον αφορά τα δεδομένα εννοούμε και αυτό θα αποσχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αθήρωση της οδηγίας ακριβώς για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα και θα κανονίσουμε μια υπουργική συνάντηση για τέτοιου είδους διαχείριση αυτών των δεδομένων του δημοσίου κατά το Συμβούλιο του Ιουνίου. Επίσης θέλουμε να υπάρξει και μια πρωτοβουλία μη νομοθετική για την τεχνητή νοημοσύνη και την ρομποτική. Θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούν ανάλογα και τα συμπέρασματα του Συμβουλίου και επίσης να τροποποιηθεί ε, σχετική νομοθεσία της Ένωσης. Ευκαιρίες και προκλήσεις υπάρχουν στο ίντερνετ και στα αυτόνομα συστήματα. η έρευνα υψηλή απόδοσης θα πρέπει επίσης να κατοχυρώσουμε την πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτούς τους τομείς και επίσης αρχάς του έτους να αναλάβουμε νομοθετικές πρωτοβουλίες για ένα οικοσύστημα ασφαλές για τις ε, ιντερνετικές πλατφόρμες και έτσι να υπάρξει η σχετική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις και για το ιντερνετικό περιεχόμενο αυτών των πλατφορμών. Πολλές χώρες υφίστανται ή τέλος πάντων εμπλέκονται σε αυτό το θέμα, οπότε θα πρέπει στο Συμβούλιο να συγκροτήσουμε κάποια προπαρασκευαστικά όργανα για αυτό το σκοπό. Τώρα για το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο του 2020 θα αρχίσουν στην Προεδρία μας οι, οι συνεννοήσεις και θέλουμε να καλύψουμε εκεί και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Οπότε θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη πρικοδότηση για χρηματοδότηση της ψηφιακής υποδομής, της ε, μεταβατικής φάσης που να περάσουν για να μετασχηματιστούν οι υπηρεσίες και η ασφάλεια. Οπότε οι ψηφιακές πολιτικές στα Δυτικά Βαλκάνια της Ένωσης θα πρέπει να προωθηθούν, να έχουμε ευρυζωνική πρόσβαση για όλους και να έχουμε συνδεσιμότητα διασυνοριακή πολύ γρήγορη και να προσέξουμε το πώς μέσω του κοινοτικού δικαίου θα επικρατήσουν, θα επικρατήσει η κατάργηση των χρεώσεων της περιαγωγής. Έχουμε Διάφορε πρωτοβουλίε που θα αναλάβουμε για όλα αυτά και όπω γνωρίζετε το σύνθημά μας για την Προεδρία μας δηλαδή είναι ο εν τη η δύναμη. και πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και σε στενή συνεργασία με εσάς θα πετύχουμε πολλά για την ενιαία ψηφιακή Ευρώπη. Οπότε σίγουρα και υπολογίζουμε στη βοήθειά σας. Και σας ευχαριστώ. Εμείς έχουμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Υπουργέ. Και τώρα. Ευχαριστώ και τους ε, κυρίους Υπουργούς. Εγώ θα αναφερθώ στα ψηφιακά και στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, στο θέμα αυτό. Έχει μεγάλη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Και εγώ νομίζω ότι έχουμε εξαιρετικούς εταίρους ε, στη Βουλγαρική Προεδρία. Υπάρχουν δύο τομείς ε, θεμελιώδες λοιπόν ε, στον ευρωπαϊκό μια προσέγγιση της χρήσης του σε όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πτυχές όπως η διάρκεια της χρήσης των αδειών κάτι που έχει τεράστιο αντίκτυπο στις επενδύσεις, καθώς μιλάμε για επενδύσεις με πολύ ψηλό κόστος. Την 1η Φεβρουαρίου θα έχουμε ένα τριμερή διάλογο, τον επόμενο τριμερή διάλογο. Εκεί πρέπει ήδη να κλείνουμε τα θέματα που αφορούν το φάσμα και φυσικά υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις, ε, πολιτικές ομάδες συμφωνούμε. Έχουμε την ίδια θέση στο θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να οφήσουμε τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο να κατανοήσουν ότι αυτό είναι αποφασιστικό. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα ακόμα στον επόμενο τριμερή διάλογο και έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο να κλείσουμε και για το έργο που συνοδεύει τη στάση αυτή. Α, μας. Εξάλλου έξι μήνες δεν είναι τραγικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την ε, αρχή με μεγάλη ταχύτητα. Εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Κορουμπάτσεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, και να σας καλωσορίσω εδώ, εξ ονόματος ε, της ε, Σοσιαλδημοκρατικής Ομάδας. Ε, αυτό είναι. Η Επιτροπή μας εδώ είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε στενά τις ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο επειδή η Βουλγαρία έχει την Προεδρία αυτή τη στιγμή. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ότι τρία πολύ σημαντικά θέματα εγκρίθηκαν στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι στόχοι του Κοινοβουλίου εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα. 35% ΑΠΕ και Βεβαίω αυτό είναι αντίθετο με αυτό το οποίο θέλει το Συμβούλιο. 30 και 27% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαι σίγουρο ότι θα γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ αυτών των στόχων. Και θα ξέρετε ότι και για αυτούς τους ε, στόχους η ομάδα μας έχει στόχο 40%. Μια άλλη ομάδα που συζητήθηκε χωρίς συνένεση ήταν οι λεγόμενοι δεσμευτικοί στόχοι για τα κράτη-μέλη. Τώρα έχουμε την εμπειρία για το πρώτο πρόγραμμα το 2020. Εκεί είχαμε δεσμευτικούς στόχους και πιστεύω ότι το πρόγραμμα αυτό έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Και βεβαίω όταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα φτάνει σε ένα σημείο, εκπληρώνει τον στόχο του. Κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν εκπληρώσει του προηγούμενους στόχους και τώρα ορίζουν νέους. Λίγο περίεργο αυτό. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και η συνδεσιμότητα. Ξέρετε ότι έχουμε φιλόδοξους στόχους για τις ΑΠΕ και αυτό οδηγεί σε τεράστια προβλήματα όσον αφορά την συνδυσιμότητα. Ο στόχος του 10% δεν έχει ακόμα επιτευχθεί και τώρα μιλάμε για ένα 15% συνδεσιμότητας. Αυτό είχε αναφερθεί στην τρίτη έκθεση περιδιακή. Βεβαίω το εάν σταματήσαμε τελείως σε ένα θέμα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει η σε όλα τα άλλα θέματα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά. Σημαίνω εδώ ότι το Nord Stream 2 δεν είναι το μόνο έργο μεταφοράς αερίου. Και τώρα απευθύνομαι στον ε, κύριο Υπουργό. Κάτι Αν καταφέρουμε να μειώσουμε βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση. Έχετε αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο. Κυρία, λοιπόν, να σας ρωτήσω το εξής. πώς θα λάβετε υπόψη την συγκεκριμένη σώτερο σε μια ενιαία προσέγγιση, συγκεντρωτική σχεδόν, για την ενέργεια. Και βεβαίως, εντάξει, η ομάδα είναι πολύ πιο ευθυγραμμισμένη, αλλά πώς θα καταλήξετε εσείς σε κάποια συνένεση στο Συμβούλιο. και με ποιον τρόπο θεωρείτε ε, ότι θα υπάρξει συνένεση. Ε, ήταν μεγάλη επιτυχία να πετύχετε κάτι τέτοιο σε έξι μήνες. Φοβάμαι ότι θα πρέπει να το περάσετε στις επόμενες προεδρίες. Η ερώτησή μου προς τον κύριο Υπουργό ακολουθεί αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πιλάρντα Δεκαστήγιο για τις τηλεπικοινωνίες. Εγώ είμαι εισηγητής για την Μπέρεκ και μαζί με τον συνάδελφο προσπαθήσαμε να έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση με συνέπεια, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε χάος για το μέλλον. Γι' αυτό θεωρώ ότι Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια, φύρα, μια χείρα φιλίας προς τα κράτη-μέλη. Κάναμε δηλαδή μια προσπάθεια να στηρίξουμε τις ε, οικονομίες ε, αυτές, εφόσον προσπαθούμε να ευθυγραμμίσουμε ακριβώ το μεγάλο αυτό τηλεπικοινωνιακό πακέτο θα λέγατε ότι υπάρχει συνένεση στο Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικό να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Μήπως ολόκληρο το πακέτο θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο θεωρείτε ότι η δική σας η Προεδρία θα το ολοκληρώσει αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ε, εξ ονόματος ε, της ΑΛΔ και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία. Και να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε τις προτεραιότητες της ε, Βουλγαρικής Προεδρίας. Όπως ανέφερε ένας συνάδελφος, <coughs> έχουμε κάποια πολύ μεγάλα θέματα που εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα στα ενεργειακά και ε, δεδομένου του εύρους ε, του πακέτου αυτού έχουμε αγχωθεί πάρα πολύ για να περάσουν όλα αυτά τα σημαντικά νομοθετήματα. Αν ε, μπορείτε, σας παρακαλώ να είστε κάπως πιο συγκεκριμένοι για όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για να δούμε πότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα όσα αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ρεαλιστικά μιλώντα λοιπόν, έχουμε, θα έλεγα, γύρω στον ένα χρόνο για να περάσουμε όλα αυτά. Ε, τότε να είστε κάπως πιο συγκεκριμένοι για το πώ μπορούμε να αναμένουμε το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων και τελικά τι στόχου έχει η Προεδρία. Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολο να κάνετε εικασίες, αλλά θα μπορούσατε να θέσετε κάποια κριτήρια για το τι θεωρείτε επιτυχία και τι θα θεωρήσετε επιτυχία να έχετε κάνει στο, μέχρι το τέλος της ε, Προεδρίας σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε τώρα στους λοιπούς ομιλητές. Θα ήθελα να μην μακρηγορήσετε τόσο. Παρακαλώ, κύριο Ζωρίνιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λαμβάνει χώρα σε ένα εξάμεινο το οποίο θα σημαδεύσει και την έναρξη της συζήτησης γιατί είναι αρκετά δύσκολη και εις βάθος να έχει ξεκαθαρισμένες τις έννοιες. Ακούσαμε να μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, άκουσα να μιλάμε και για συνοχή. Η συνοχή είναι πολύ σημαντική, σημαίνει τη μείωση των ανισοτήτων. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το νέο στάδιο να εισαγάγουμε την έννοια της σύγκλησης με έναν πιο βαθύ τρόπο. Δεν μιλάμε για μεταφορά από τους φτωχότερους στους πλουσιότερους, μιλάμε για συνέργεια. Οι χώρες με μεγαλύτερη δυναμική μεγενθύνονται αυτή τη στιγμή και ε, δημιουργούν θέσεις εργασίας ε, και πλούτο όμως θα πρέπει να δημιουργήσουν θέσει εργασίας και πλούτο και οι χώρε που έχουν μικρότερη δυναμική αυτή τη φορά. Ε, αυτό ενισχύει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς σκέφτεστε να θέσετε σε εφαρμογή τους μεγάλους φακέλους της Προεδρίας σας, το φάκελο της καθαρής ενέργειας που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, το φάκελο της ευφύους κινητικότητας, ε, ε, το οποίο έρχεται να συναντήσει ε, την καθαρή ενέργεια και την ψηφιακή επανάσταση, το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων, και το θέμα των νέων. Πώς ε, θα θέσετε σε εφαρμογή λοιπόν τους φακέλους αυτούς, με ποια χρονοδιαγράμματα και πώς σκοπεύετε να θέσετε το θέμα, την αρχή της σύγκλησης ως ε, βάση υλοποίησης των πολιτικών αυτών. Γιατί η σύγκληση μας επιτρέπει ε, να έχουμε απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Έχουμε τις ευρωεκλογέ το Μέιο του 2019. Τότε αλλά και σήμερα θα πρέπει να έχουμε περισσότερα πράγματα, δηλαδή κάτι συγκεκριμένο να παρουσιάσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μοτσκόφσκι, κυρία Πέτκοβα, θα ήθελα να σας καλωσορίσω, αλλά και στον ψηφιακό. Η Βουλγαρική Προεδρία έχει αναπτύξει τις προτεραιότητές της βάση ε, των, οδών αλλά και των πηγών εφοδιασμού έχει καταστεί η προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Και θέλω να ρωτήσω το εξής ε, αερίου στα Βαλκάνια και χαίρομαι που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή οι διασυνδέσεις. Πολλοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι... Και η ερώτησή μου είναι... Στις περισσότερες από αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τίποτα δεν έχει υποθεί. Όμως, προκειμένου να εγγυηθούμε την ψηφιακή ασφάλεια, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις υποδόμες του και τους ε, δύο υπουργούς ε, που ήταν στην Επιτροπή μας. Ε, θέλω να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Πετκόβα καταρχήν για τα συμπεράσματα του βασίζεται ε, ιδιαίτερα σε αυτά τα συμπεράσματα έχουν περάσει 3,5 χρόνια από τότε. Με όρους ε, μετάβασης ενέργειας Οκτώβριος του 2014 είναι ο προηγούμενος αιώνας. Μόλις ε, πέρσι μειώθηκε μέσα. Ε, πολλά έχουν συμβεί από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τώρα, όμως το Συμβούλιο βασίζεται σε αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ιδιαίτερα λεπτομερώς. Δεν πιστεύετε ότι τη σήμερα ημέρα είναι παροχημένα αυτά τα συμπεράσματα και, το ποσοστό, και σε ποσοστό του ΕΕΠ τέσσερις φορές περισσότερο. Πιστεύετε μήπως ότι όχι και ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχος που έχει τεθεί από το Συμβούλιο θα ξαναφέρει την Ευρώπη σε ηγετική θέση ή θεωρείτε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να μετακινηθεί προς τη φιλοδοξία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς με τις δικές σας παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι, είναι πάρα πολύ σημαντικός για την οικονομία, για τους Ευρωπαίους, επικοινωνία με το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε σύγκληση απόψεων, ούτως ώστε να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα για επικοινωνία με το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να έχουμε σύγκληση απόψεων, ούτω ώστε να πετύχουμε όσο γίνεται περισσότερα για όλους τους Ευρωπαίους. Πιο συγκεκριμένα τώρα, Όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα ή του στόχου κλπ. κλπ. Πάρα πολύ σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουμε του τεμνέ διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Και στα πλαίσια αυτών των τριμερών διαλόγων η Προεδρία μα πρόκειται να απασχίσει να επιτυχούμε κάποιο είδου σύγκληση αλλά και κάποιο είδου ε, πρόοδο για όλα τα θέματα αυτά. Και πρώτα πρώτα Ερωτήσεις κ. Τωσανόφσκι, Κουρουμπάσεφ, Πέτερσεν. Για αυτά που ρωτήσατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στόχους επιτεύξιμους και λογικούς. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Ρωτήσατε κάτι είπατε για τις ιδιορυθμίες, ιδιοτυπίες κάθε κράτος μέλος. Ε, φυσικά και έχει το κάθε κράτος τις ιδιωτερότητές τους και πιστεύουμε ότι η Ενεργειακή Ένωση θα είναι βιώσιμη μόνο να λάβει υπόψη το ενεργειακό μείγμα κάθε κράτος μέλος. Τώρα, για τον κύριο Ουρούτσεφ. για συστημική διασυνδεσιμότητα στην ε, νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ναι, είναι πολύ σοβαρό και σχετίζεται με την ασφάλεια αυτής της περιοχής. Σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητά της επίσης. Το Ανατολική Ευρώπη, ναι, είναι πολύ σοβαρό και σχετίζεται με την ασφάλεια αυτής της περιοχής. Σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητά της επίσης αναπτύχθηκε, προχώρησε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε διαφοροποίηση όσον αφορά το ότι ονομάζεται Βαλκάνια αυτός ο κόμβος. Έτσι, με αυτόν τον κόμβο θα υπάρξει όθηση για την ε, εξασφάλιση της πρόκειται για τη γεωγραφική θέση της Βουλγαρίας. Ε, αυτός είναι ο λόγος. Βρίσκεται επομένως σε κομική θέση όσον αφορά τη διαδρομή αυτή. Αλλά βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο την Βουλγαρία, αφορά όλους τους Ευρωπαίους ως έργο, ως σχέδιο. Τώρα ο κύριος Πέτερσεν. Ήθελα να σας πω πιο συγκεκριμένα δύο λόγια για κάποια χρονοδιαγράμματα και για το πώς θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά την πρώτη δέσμη μέτρων που είναι πάρα πολύ σημαντική, περιλαμβάνει τον κανονισμό για την διακυβέρνηση, την οδηγία για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και για αυτή τη θέση μέτρων θα αρχίσουμε κατά τα τέλη του μηνό ε, τον διάλογο με το Κοινοβούλιο μέσω τρίμου διαλόγου. Και πιστεύουμε πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο. Να πετύχουμε έτσι μια συνένεση. Οπότε να έχουμε κοινή προσέγγιση και για έναν άλλο πάρα πολύ σημαντικό οργανισμό αυτόν που ονομάζεται Acer. Και βασική μας προσέγγιση και στόχος είναι να συνεχιστεί αυτή η θετική τάση στις επαφές, στις συζητήσεις και να συνεχίσουμε την οριζόντια προσέγγιση μια που καθένα από αυτά τα θέματα είναι, είναι συγκεκριμένα αλλά όλα έχουν συγκεκριμένο ρόλο λειτουργία ε, στο όλο πακέτο, στην όλη δέσμη. Σας ευχαριστώ την προσοχή σας. Αν θέλετε μπορείτε και αργότερα να απαντήσετε σε κάτι, αλλά τώρα να... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο στόχος μας είναι να αναπτύξουμε έξυπνο δίκτυο, την πέμπτη γενιά τηλεφωνίας, αυτόνομα αυτοκίνητα και να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη που έχουμε και να συνεργαστούμε. Να συγχρονίσουμε τις ε, δράσεις μας Δυστυχώς για να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα γιατί υπάρχουν κάποιοι πόροι ανεκμετάλλευτοι για την τέταρτη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται γρήγορες και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ακριβώ τα θέματα υποδομών για να έχουμε επαρκή Οπότε θα προσπαθήσουμε να οριστικοποιήσουμε την αναθέτηση για τις ε, χρεώσεις ε, περιαγωγής ε, τρίτες χώρες να γίνει από την σκόπια της Προεδρίας ε, και σε συμφωνία με όλα τα θεσμικά. Είναι θετικό το ότι του ενός λεπτού ομιλίας από την Πουδουμού στην Σερβία είναι 4 ευρώ, δηλαδή τεράστιο ποσό για δύο χώρε γειτονικέ ε, εφαρμογές όταν ο κόσμος κάνει τουρισμό ή πάει για δουλειά να μπορεί να έχει φυσιολογικές τιμέ ε, για το Τώρα για την ερώτηση του κυρίου Ζουρινιά. βήμα έτσι ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή ψηφιακών πρωτοβουλειών, να εναρμονίσουμε περισσότερο τις προδιαγραφές. Είναι πράγματα πολύ σημαντικά για την ψηφιακή μετάβαση. Την ε, κυβερνοασφάλεια. της ε, κυβερνάλειας. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα βασικό επίπεδο ασφαλής, το οποίο θα συνεισφέρει. Και θα απαιτηθεί και κάποια πιστοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν. περισσότερη προσπάθεια. Ο πρόεδρος. Έχουμε ακόμα 4-5 λεπτάκια. Οπότε αν κάποιος έχει κάποια ερώτηση. Κύριε Τούρμες. Ήμουν ασκιώδης ε, εισηγητής ε, για το market design. Εσύ ε, ότι θέλετε να δείτε και μια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πέρα από τα σύνορα στα Βαλκάνια και πέρα στην Ευρώπη. Να δούμε λοιπόν ότι για τον επόμενο 1,5 χρόνο με τη Βουλγαρική, Αυστριακή, Ρουμανική Προεδρία έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε στις Βαλτικής. Έτσι λοιπόν, αν ε, μπορείτε μια μελέτη για την ε, Ευρώπη και κάτι που με εξέπληξε ήταν ότι η Βουλγαρία μαζί με την Πορτογαλία και μαζί με ένα τμήμα της Ισπανίας έχει ε, τον πιο αποδοτικό προς το κόστος δυναμικό κατάσταση λόγω του δεσμευτικού στόχου του 2020 το Λουξεμβουργό θα πρέπει να αγοράσει στατιστικές ε, μεταφορές, η Γαλλία, οι κάτω χώρες θα πρέπει να αγοράσουν. Γιατί λοιπόν η Βουλγαρία δεν ε, βλέπει την ευκαιρία αυτή να, να μεταφέρετε την ενέργεια αυτή, να τη μεταβάσετε και να πληρωθείτε. Γιατί ε, τελικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Βουλγαρία μπορεί να είναι ένας μεγάλος νικητής από μια ε, ταχεία μεταβίβαση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνω, η ερώτηση αφορά την ε, κυρία Πέτκοβα που είναι αρμόδια για την ενέργεια, για τις ενεργειακές αγορές. Φυσικά, το ψηφιακό θεματολόγιο είναι πολύ σημαντικό για τα... στην ερώτηση αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Τούρμες, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανανεώσιμε πηγέ. Ο στόχος μας είναι 16% μέχρι το 2020. Και εμείς έχουμε υλοποιήσει το στόχο αυτό ήδη από τα τέλη του 2014 και στα πλαίσια της Βουλγαρικής Προεδρίας θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που κατέχουμε σε όλες τις συζητήσεις. Ότι αυτό είναι ένα περαιτέρω βήμα που σκοπεύουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από ό,τι βλέπω. Από το κρατήριο σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο. Σάμινο και πάλι σας ευχαριστούμε. Και τώρα... Θέλουμε να καλωσορίσουμε δύο ακόμη υπουργού. Uh, well, uh, next ministers in front of us, uh, of the Council. Κασιμίρ Βάλτσεφ, Υπουργός Παιδείας και Επιστημών. Θα ζητήσω και από τους υπουργού, να πάρουν το λόγο. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, να παρουσιάσω εκ νέου. Καλωσορίζω και τους δυο σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Υπουργό Καρανικολόφ, ο οποίος είναι υπουργός Οικονομίας, για μας σημαίνει για τη βιομηχανία και να καλωσορίσω και τον κύριο Βάλτσεφ, ο οποίο είναι υπουργό Παιδεία και Επιστημών από τη δική μα σκοπιά. Είναι αρμόδιο για το θέμα τη έρευνα. πολύ σημαντικό. Να λάβετε το λόγο για μια εισαγωγή 7-10 λεπτών. Καταρχήν το λόγο έχει ο κύριος Καρανικόλοφ και κατόπιν ο κύριος Βάλτσεφ και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Καρανικόλοφ, καταρχήν. Κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες μας γιατί έχουμε μία θετική εξέλιξη στη βιομηχανική μας πολιτική. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει μια συνέχεια, θα πρέπει να συνεχίσουμε τα όσα σωστά έχουν γίνει από πλευρά ε, Τρόικα, αλλά και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2017. Οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ετών αλλά και κάποια συστηματικά προβλήματα ε, είναι αποτέλεσμα της κρίσης, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους μακρόπνο πλαίσιο για την βιομηχανική. Αμοιές μας έχουν πολλές ε, προκλήσεις, οπότε έχουμε εξέλιξη την τεχνολογία, άρα αλλάζει και η οικονομία. Και οι φραγμοί που απομένουν ε, στο δρόμο της βιομηχανίας μας ε, σημαίνουν ότι θα πρέπει να δουλέψουμε εντατικά σε αυτή την κρίσιμη καμπή την Προεδρία. Ήρθε η ώρα ούτω ώστε η ολοκλήρωση ε, η Ευρωπαϊκή να τονωθεί, να αναβαθμιστεί. Οι έξι δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η έχει πετύχει και να πετύχει περισσότερα με κοινέ λύσεις οι οποίες ε, μπορούν να ωφελήσουν την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με ρεαλισμό, έχοντας επίγνωση των ε, εκτιμάτων μας και εκτιμάτων μας και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ξέρουμε ότι εσείς είστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων. Και θα πρετανεύσει το πνεύμα της συνέχειας, γιατί αυτό θα πει προϋπόθεση επιτυχίας, δηλαδή μια κοινή προσπάθεια. Και είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, το οποίο είναι ευχάριστο, γιατί έχετε κάνει πολλά για την ε, ανάπτυξη, και τη χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής. Από πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οπότε αυτή η συνολική ανακοίνωση που αφορά σφαιρικά τη βιομηχανική πολιτική και καλύπτονται όλες οι μέρους πολιτικές που αποσκοπούν στην ε, ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Άρα θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την προσέγγιση, θα πρέπει να υπάρχει λύση για να μπορέσει να συνεχίσει να ανταγωνιστική η Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή πολιτική που να αφορά στενό συντονισμό Ευρώπης κρατών μελών και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιου είδου κοινού στόχους. Να ελκύσουμε επενδύσεις χρειάζονται μακροπρόθεσμοι ε, στοιχεία προβλεψιμότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης οι παγκόσμιοι εταίροι αλλά και οι ανταγωνιστές μας ήδη έχουν τέτοιου είδους μακρόπνες ε, και για την ε, καινοτομία. Έτσι θα έχουμε προσθεμένη αξία. Αν έχουμε κάποιους τομείς ε, έντασης γνώσης, έτσι θα στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα, θα την εξελίξουμε και χρειαζόμαστε τις επενδύσεις και την καινοτομία και σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους του ώστε οι πιο ταλαντούχοι να μείνουν στην Ευρώπη ανάπτυξη και ευημερία χρειάζονται εάν εμβαθύνουμε στην ενιαία αγορά να μην υπάρχουν φραγμοί για τις επιχειρήσεις, χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην αγορά των τρίτων χωρών θα πρέπει η επαγγελματική κατάρτιση και η Αν έχουμε επενδύσεις σε τεχνολογίες ήταν πολύ θετικό. Το ε, βιομηχανία 4-0. Και έχουμε το Συμβούλιο Ανταγωνισμού και Ανταγωνιστικότητας ε, όπου θα πρέπει να αποφύγει πιο συγκεκριμένα θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Το Συμβούλιο θεωρεί είναι πάρα πολύ θετική. Περισσότερα κίνητρα για αυτές τις ε, ε, μη και τις κελάψης ούτω ώστε να φτάσουμε σε κάποιο είδου την αποτελεσματικότητα του προγράμματο και τα αποτελέσματά του. Οπότε και από κοντά θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη ε, τη διαστημική πολιτική, να δούμε τι θα γίνει με το Κοπέρνικο. Μάρτιο βασικά θέματα εκεί θα είναι το πώς ο διαστημικός τομέας θα είναι ανταγωνιστικός ε, παγκοσμίω και πώς διαπραγματεύσεις που αφορούν την ε, αμυντική μας βιομηχανία και θέλουμε αυτό να γίνει όσο γίνεται συντομότερα για έκαναν για την αξιολόγηση του ορίζοντα 2020 και του προγράμματος πλαισίου 9 που ορίζει ξεκάθαρα την δυνατότητα χρήσης ε, της ε, σύνδεξης ε, για το καλό της ανθρωπότητας. Το ITER είναι ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας για το μέλλον τη ανθρωπότητας και συνεργάζεται εκεί πέρα Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Νότια Κορέα και ΙΠΑ κάτω του νέου Προέδρου του ΙΤΕΡ, του καθηγητή ε, Μπίγκο, για να ε, έχουμε μια διαχείριση του κόστους. Αναμένω βεβαίως την ίδια στήριξη και από το Συμβούλιο όταν μιλάμε για την έγκριση από την ε, Κίνα, Ιαπωνία, ΙΠΑ και αλλού. Είναι λοιπόν ε, πάρα πολύ σημαντικό να επεκτείνουμε το ευθύναμε λοιπόν έτοιμα στην Επιτροπή σας να υπάρξει κάποια γνωμοδότηση για το ΕΒΡΑΤΟΜ Η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει μια σειρά σημαντικών φόρα για την έρευνα και την καινοτομία και θα ήθελα να έχουν ευκαιρία να σας καλωσορίσω για το πώς θα μπορέσουμε ε, για, το, για τη συμμετοχή του στην Σόφια στις 25 ε, και 26 Μαρτίου για την ερευνητική υποδομή αλλά και για το μέλλον ε, των τροφίμων, της υγιεινής διατροφής ε, και των 25 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τους υπουργούς. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Ο κύριος Έλε. Ευχαριστώ και τους υπουργούς. Έχω μια ερώτηση για το πρόγραμμα πλαίσιο και την καινοτομία για τον κύριο Βάλτσεφ. Εκτιμούμε την Βουλγαρική Προεδρία γιατί πιστεύουμε ότι είναι ε, πολύ σημαντικό και πήγον ε, πριν ε, από το πρόγραμμα να κάνουμε μια συζήτηση για το χάσμα καινοτομίας στην Ευρώπη. Αλλά εδώ και 15 χρόνια εγώ ε, προωθώ το να διευρύνουμε τα μέσα. Θα πρότεινα να ρίξετε μία ματιά στη μελέτη που κάναμε για τη ΣΤΟΑ για το χάσμα στην καινοτομία. Πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό, αν θέλετε να το πετύχετε αυτό, ε, σαν ε, να πάρετε ε, τη θέση των ψευτών, το χάρη, αυτών που κάνουν μπλοφαρούν στο πόκερ. Ε, χάρη χάρη, όμω δεν αντιμετωπίστηκε το ζήτημα. Και θέλω να ρωτήσω. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η Κομισιόν δίσταζε για το θέμα αυτό, γιατί σε κάποιο βαθμό εντάστηκε στις αρμοδιότητες των κρατών μελών το πρόγραμμα να ε, έχει να κάνει με προγράμματα μεταρρυθμίσεων ε, στο πλαίσιο των υποδομών. Και θα ήθελα να πω σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτό. Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η αριστεία δεν έχει να κάνει μόνο με την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά σχετίζεται και με διευθυντικές ικανότητες, ε, σχετίζεται και με τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε σκηνοπραξία. Ένα κράτος μέλος ε, ήθελε να έχει ένα πρόγραμμα αριστείας, αλλά ε, η αναφορά θα ήταν ευρωπαϊκή, αλλά στη συνέχεια θα έδινε χρήματα σε ε, θεσμούς που θα είχαν επιλογή και, επιλεγεί και απευθείας από το πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό και για μια θεσμική αλλαγή, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη νεότερη γενιά κτλ. Δηλαδή, για μια χώρα σαν την Βουλγαρία, για μια μεγάλη χώρα, μήπως ε, σκέφτεται να αναλάβει μια ηγετική θέση σε μια τέτοια συζήτηση για το ε, ποια εργαλεία θα έπρεπε να έχει το πρόγραμμα που γίνονται στις ίδιες χώρες σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και για τις παρατηρήσεις σας, ο κύριος Μαρτά, για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Είμαι ο τελευταίος ε, που παραμένει. Δεν ξέρω τώρα αν ε, οι υπόλοιποι της ομάδας ε, θα συμφωνήσουν με αυτά που λέω. Για την Βουλγαρία έχουμε τώρα μεγάλη πρόκληση την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπατε κύριε Υπουργέ Οικονομίας θα εργαστείτε για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα ε, της οικονομίας. Αυτό το κοινοβούλιο έχει εργαστεί το 2016 και το 2017 ε, γύρω από το θέμα της οικονομίας της αγοράς, ε, το καθόδες των χωρών, ξέρετε την Κίνα κτλ. Έτσι λοιπόν θα σας ξαναθέσω την ερώτηση που έθεσα και στους συναδέλφους που έφυγαν μόλις. Ελπίζω να μπορέσετε να μου απαντήσετε. Ταυτόχρονα, ε, όπως σας είπα, είναι μεγάλο το έτος γιατί η Βουλγαρία θα μπει και στην ομάδα των 16 συν 1 ε, και τι ακριβώς θα γίνει ε, με τις κινέζικες επενδύσεις στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακάπτοντας τους κανόνες Ευρωπαϊκή Ένωση, και ξέρετε ότι αναφέρομαι σε δρομική γραμμή Βουδαπέστη ε, Βελιγράδη και στα πλαίσια του 16 στην 1 έχετε υπογράψει μια συμφωνία με την Κίνα για ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό ουσιαστικά ε, αντιτίθεται στην δουλειά που έχουμε κάνει προκειμένου να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας έτσι ώστε να μπορούν όλοι να δρούν με ίσους κανόνες. Ε, δηλαδή αυτή η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών αντιτίθεται σε αυτά που κάναμε. Και ξέρετε ότι και η Κομισιόν δικαίως ανησυχεί για τις ξένες επενδύσεις και ε, ουσιαστικά προβαίνει σε μία επιχείρηση ε, εποπτείας ε, αυτών των ε, επενδύσεων σε τομείς ευαίσθητους όπως οι μεταφορές, ψηφιακή οικονομία κτλ. Η ερώτηση λοιπόν που σας θέτω είναι ποια θα είναι η στάση σας στο εξάμενο αυτό ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι η Κομισιόν σε εισαγωγικά μπορεί να εργαστεί κατά των συμφερόντων της χώρας σας και της ομάδας 16 1. Δηλαδή, είναι κάπως ε, αντιφατική η πραγματικότητα αυτής της ομάδας 16 συν 1 και να λειτουργείται στα πλαίσια αυτής της ομάδας. Ερώτησή Η πολιτική συζήτηση για τις επενδύσεις ε, στην έρευνα και το εάν ε, πρέπει να κατευθύνονται προς την αριστεία ή προς τους υπουργούς Αυτές οι συζητήσεις γίνονται και στις ε, δικές τους ε, χώρες. Ε, είμαι σίγουρος πως θα έχουμε την δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να γίνει πιο περιληπτικό και να περιλαμβάνει και άλλες χώρες να σπάσουν οι κλειστές ε, λέσχες ε, και να μπορούν να ενταχθούν και άλλοι συμμετέχοντες. Ας ε, περιμένουμε να δούμε τι θα μας προτείνει η Κομισιόν τον Ιούνιο. από το πρόγραμμα πλαίσιο και θα προσπαθήσουμε ακριβώς να δημιουργήσουμε συνέργειες για να υπάρχουν ουσιαστικότερα αποτελέσματα στην κοινωνία και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τα Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, εμείς επενδύουμε στην ερευνητική υποδομή, οικοδομούμε έργα αριστείας και σκοπεύουμε ε, να δημιουργήσουμε και περιφερειακές υποδομές. Για εμένα είναι σημαντικό να προωθήσω την αριστεία και την ε, εκπαίδευση σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την έρευνα αυτή, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να αντλήσουμε γνώση για το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, ε, τις ομιλίες σας και τις απαντήσεις σά λοιπόν, Σας ευχαριστώ, ποιητή Υπουργή, για την παρουσία σας, ε, τις ομιλίες σας και απαντήσαμε στα ερωτήματα βιομηχανία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καινοτομία, ε, διάστημα και έρευνα. Αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν όλο το εξάμεινο. Πολύ σημαντικό εξάμεινο, το τελευταίο εξάμεινο δώσουμε το έργο μας. Οπότε είναι απολύτως αναγκαίο να προχωρήσουμε τόσο το μοτρό δυνατόν. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και πύλη. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Κανονισμός ε, της ε, Κομισιόν 347 του 2013 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος λοιπόν. Καλώς ορίζω την κυρία Κατερίνα Σίκοφ, ε, προϊσταμένη της αρμόδιας μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Θα θέλαμε λοιπόν να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά μαζί σας. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόσκληση της Επιτροπής μας για να μας παρουσιάσετε την ε, πράξη κατεξιοδότηση για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος ε, που έγιναν σύμφωνα με τις κατακτήριες γραμμές. Έργα κοινού ενδιαφέροντος. Είναι έργα υποδομών, ειδικά διασυνοριακά έργα που διασυνδέουν τα ενεργειακά συστήματα των κρατών μελών. Στόχο έχουν να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους ε, που αφορούν την ενέργεια και το κλίμα και να απομακρυνθούμε από τις εκπομπές άνθρακα κάθε δύο χρόνια η Κομισιόν ε, συντάσσει ένα νέο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος. Καλώς ήρθατε κυρία μου. Έχουμε λοιπόν την εξέταση εδώ των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της ε, Κομισιόν. Η πράξη αυτή κατεξιοδότηση μας διαβίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. Ζητήσαμε παράταση της δίμηνης ε, περίοδου για να αξιολογήσουμε σωστά την πράξη αυτή κατεξιοδότηση Οπότε 27 Μαρτίου ολοκληρώνεται η περίοδος. Επίσης, να πω αγαπητοί φίλοι κάτι το πολύ σημαντικό, η προθεσμία για αντιρρήσεις από τα μέλη της Επιτροπής μας είναι η 26 Ιανουαρίου 2018 στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τη στιγμή εκείνη λοιπόν μπορεί να πούμε αντιρρήσεις ε, για την πράξη αυτή κατά εξουσιοδότηση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε, αγαπητή μου κυρία. Και το θέμα βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Πάμε προς τα μπρος. Ήδη, ήδη είδαμε την ε, πρώτη επιτυχία της εφαρμογής ε, της πολιτικής αυτής και στην περίπτωση αυτή, τα περισσότερα κράτη-μέλη, 24 κράτη-μέλη, πιθανές διακοπές του φωδιασμού. Για την ηλεκτρική ενέργεια οι προκλήσεις μεγενθύνονται αντιθέτως. Να πάρει την παραγωγή ενέργειας από νέες πηγές, από εκεί που παράγεται, και όπου χρειάζεται και στα νοικοκυριά τον ηλεκτρισμό. Βλέπουμε στο αέριο κάποια project που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο και ε, φυσικά κάποιο θα καταστήσεις ε, στο περιβάλλον και δεν δοθεί η άδεια, εντάξει. Έτσι, λοιπόν, ε, αυτή η άδεια, ο κατάλογος των έργων αυτών, δεν ε, αφορά επιδοτήσεις για έργα. Ε, περιμένουμε μέσω των επιδομάτων για έργα ή μέσω του σχεδίου Juncker θα δεχθούν χρηματοδότηση, μόχλευση, χωρίς να υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση και το τρίτο, στην Βαλτική, στην ε, Βουλγαρία, στην Πολωνία κτλ. Αυτό γιατί τα project του αερίου τα έχουμε προετοιμάσει. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσία στη συζήτηση αυτή και ελπίζω ότι με την ευκαιρία αυτή και η Κομισιόν κατά νου. Για να είμαστε συνεκτικοί, πιστεύω ότι θα ήταν καλό η συζήτηση αυτή και μάλιστα για να καταλάβουμε και ποιος είναι ο βαθμός ε, ε, ουσιαστικά πλήρωσης κάποιων δικτών. Μιλήσατε για, για Αυστρία, Τσεχία, ε, όπου έχουμε ένα πολύ σκληρό χειμώνα και αν ε, για έξι ώρες ε, δεν έχεις θέρμανση τότε είναι αλωσή ανθρακά. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν λύσεις για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της λειτουργίας των ενεργειακών προβλήματα. Και τότε το χάρη, όπως ε, γίνεται με τον αγωγό που υπάρχει μεταξύ Βουλγαρίας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας. Ε, με ένα πολύ πιο σοβαρό τρόπο, γιατί δυστυχώ η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνούμε ή διαφωνούμε, είναι θέμα επιβίωσης ε, για του πολίτε μα. Αυτή καταρτήσουμε από κοινού αυτέ τι λίστε έργων κοινού ενδιαφέροντο και θα κάνω και ένα σχόλιο. Αλλακτικέ ΑΒΓ. Συγγνώμη που θέτω τέτοιε ερωτήσει, αλλά αν είχαν γίνει συζητήσει εκ των προτέρων, ε, μάλλον δεν θα χρειαζόταν να κάνω και αυτέ τι ερωτήσει. Πάντω σα ευχαριστώ. Δεν με είδατε καλά, τι να εδώ, εδώ στα, στα, ε, Είναι σύντομο. θα είναι στο ίδιο μήκο κύματο αυτό ο καταλόγο. Δεν ισχύει όμω αυτό. Μα τι είναι αυτό, είναι αυτό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Πού το, είναι μήπως ε, αριστερή, ε, είναι μήπως ε, οικολόγος, όχι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα όλα αυτά τα... Και νομίζω ότι αυτή η επιλογή θα έπρεπε να είναι στο ίδιο μικρό σχήματος με τους στόχους που θέσαμε και το COP21. Θα σίγουρα θα ξέρετε ότι θα έχουμε από το φράκινγκ φυσκόρη από την Αλγερία. Μπείτε στη θέση των Ευρωπαίων. Δεν πρόκειται να καταλάβουν με τίποτα. Μπορούν να χωνέψουν πώς φτιάξατε αυτήν την λίστα, αυτόν τον κατάλογο. Μα θα πρέπει να ρωτήσετε τους ερετούς άρχοντες, τους ντόπιου, τον κόσμο να διαβολευτείτε. Άρα θα πρέπει να, δούμε από... Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κάποιο άλλο τον λόγο. Από το κέντρο, εκεί στα δεξιά. Δεν βλέπω σωστά τα πράγματα από πάνω και νομίζω πως η συζήτηση η κανονική συνεπτοπή μας θα είναι κάπως ε, διαφορετική, αλλά τώρα είμαστε στην αρχή και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τις απαντήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλια. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες, αλλά ίσως κάποιες μπορούν να απαντήσουν με κάποια πιο γενικά σχόλια. Να ξεκινήσω με αυτό λοιπόν. Πρώτα απ' όλα η ανάλυση έγινε με το σενάριο ότι οι στόχοι για τις ΑΠΕ και το κλίμα θα επιτευχθούν για το 2020. Δηλαδή οι αναλύσεις που κάνουμε οπότε οι στόχοι ενεργειακής αποδοτικότητας ε, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, εκπληρώνονται και υποθέτουμε επίσης ότι θα έχουμε και τη σχετική νομοθεσία και μάλιστα νωρίς και όχι αργά. Όλα αυτά είναι ένα σενάριο. Κάναμε την αξιολόγηση των αναγκών αφορούν τους τρεις πυλώνες της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα δηλαδή η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς όπου εξετάζουμε το τι τιμές πληρώνουν οι πολίτες για αέριο και ηλεκτρικές τιμές από ό,τι αλλού στην Ευρώπη, τότε λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ανταγωνισμός, ανταγωνισμός ο οποίος μετά μειώνει και έτσι μπόρεσε να εξοφλήσει τον σταθμό κλαϊπέντα σε δύο χρόνια παρόμοια Ευρώπη έχει πρόσβαση σε ανταγωνιστικές τιμές, τότε η οικονομία είναι της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ηλεκτρισμού και αερίου. Αυτές είναι λοιπόν οι διαφορές αερίου που βλέπουμε στην εσωτερική αγορά, ειδικά στο αέριο. Η εφοδιαστική ασφάλεια σημαίνει ότι υπάρχουν εναλλακτικές οι οποίες μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν ή θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθούν εκτός το αέριο είναι ότι το δίκτυο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2020, ενώ στον ηλεκτρισμό οι ανάγκες αυξάνονται. Να φερθώ και στις λεπτομέρειες. Βεβαίως δεν μπορώ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο διάλογος που κάνουμε είναι με ενδιαφερόμενος ε, και 21. Όπως είπα, εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2030 σε ανα πάσα στιγμή. Λαμβάνοντας υπόψη ε, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ για να πετύχουμε τους στόχους ε, του 30% ως μέρος της ανάλυσης κόστους οφέλους έχουμε δει τον αντίκτυπο που υπάρχει στο περιβάλλον. Γι' αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω ότι είχαμε μια συνεπή προσέγγιση και πάντα υπάρχει ομαδοποίηση. Αλλά είναι, γι' αυτό είναι και δύσκολο τι πρέπει να γίνει στην Ευρώπη. Και συνένεση στο ότι πρέπει η προτεραιότητα να δοθεί στον ηλεκτρισμό. στα ανταγωνιστικά έργα. Μιλάμε για το πώς θα έχουμε αέριο στην αγορά και κατά κανόνα ένα έργο υπάρχει αλλά θα ξαναδώ, κατά κανόνα βλέπουμε τον κατάλογο κάθε δύο χρόνια και αν το κόστος αυξηθεί, παραδείγματος χάρη, θα επανεξτάσουμε τα έργα, γιατί είναι σχεδόν αδύνατο και ίσως ε, το έργο πλέον να μην είναι βιώσιμο από κοινωνική σκοπιά. Έχουν διάρκεια ζωής 20 έως 40 και σε ορισμένες περιπτώσεις 60 έτη. Είναι γεγονός. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να αξιολογήσει η αγορά και αναμένουμε ότι η αγορά σε περισσότερες περιπτώσεις ε, θα πιστεύουν ότι το χρειάζονται για τα επόμενα 10 χρόνια ή 20 χρόνια θα το κάνουν. Εάν θεωρούν ότι θα πρέπει να κάνουν απόσβεση σε 40 χρόνια, μάλλον θα αναρωτηθούν εάν αξίζει τον κόπο. για το σχόλιο περί εταιρικών συμφωνίου και βεβαίως μας έχουν οι ρυθμιστικές αρχές μεταξύ των οποίων και η υπηρεσία Acer και η Κομισιόν και οι περιφερειακές ομάδες. Οπότε δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Δεν έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα που αφορά εταιρικά συμφέροντα. όσον αφορά τους διαχειριστές του δικτύου μετάδοσης. Κατόπιν, για να ολοκληρώσω, όλες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές είναι μέλη του δικτύου μας. Πολύ σημαντικά μέλη, γιατί αυτοί λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό συμφέρον και είναι ευθυγραμμισμένοι ευθυγραμμισμένοι δρομενές υπηρεσίες. Έχουμε αυτή την περιφερειακή συνεργασία και ίσως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου κάποια έργα μπορεί να μην ωφελήσουν μια χώρα, αλλά ωφελούν τη γειτονική χώρα. Αυτό εξετάζουμε την ευρωπαϊκή σκοπιά. Οπότε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι εντός αυτού του πλαισίου για την ε, χρηματοδότηση. Έχουμε την διαδικασία προγραμματισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την περιφερειακή συνεργασία και την εμπλοκή των ρυθμιστικών αρχών. Η δρομία ως πολιτικός. Γιατί θα πρέπει να είμαστε μετριοπαθείς ως πολιτικοί αν θέλουμε να πετύχουμε το οτιδήποτε. Έχουμε ακόμη λίγα λεπτά. Θα έχουμε ένα δεύτερο μέρος δεν έχει τελειώσει. Όχι, όχι. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας. Ε, θα έχουμε ένα δεύτερο μέρος. Δεν έχει τελειώσει. Όχι, όχι. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας. Πρέπει να πάω στον Επιτροπή Επασχόλησης, λέει ο κ. Μαρτά. Κρίμα. Το σημαντικό μέρος τώρα ξεκινάει. Äh, Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίαση. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον για το Κοινοβούλιο να βλέπουμε που δίνεται βάρος, ειδικά στην τόρινη συγκυρία που πρέπει να βλέπουμε ακριβώς ε, το πώς ε, θα εξελιχθεί Εκεί πέρα υποθέτουμε ότι θα έχουμε κάποια ισότητα στο, των εντός και των εκτός και βέβαια να έχει σημασία και η ενεργειακή χάρτα η οποία έχει τέτοια μορφή ώστε όλα τα μέρη να έχουν μια ευρωπαϊκό επίπεδο να το λαμβάνουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ε, δείτε τα πρώτα έργα που είχαν ξεκινήσει πριν από μία δεκαετία. Να δούμε και τη διαφορά μεταξύ διαφόρων ε, κλάδων, ε, ρεύματος και αερίου. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις... Όσο υπήρχε αμερικανική παραγωγή εντωμεταξύ χρεοκόπησαν 6.000 εταιρείες γιατί ποια είναι τα κενά στο γράφημά σας ότι είναι δηλαδή ε, προς το κοινό συμφέρον είναι αναμφισβήτητο. Αλλά δυσκολότερα είναι τα πράγματα στην αγορά του ρεύματο. Δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε εκεί όπου χρειάζεται, ώστε η Γερμανία πριν από 10 μέρες πλήρωσε την Ολλανδία για να πάρει ε, να δούμε και τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του αερίου που δεν υπάρχουν στον καταλογό σας όπως το... Πιο Ευχαριστώ. Να Προτείνω τον κύριο Μπενίτο Σιλουάγα ως τελευταίο μιλητή. Τι απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, η συζήτηση και σίγουρα θα είναι πολύ ικανοποιημένο ε, να συζητήσει μαζί σας ε, πολύ πιο έγκαιρα στη διαδικασία. Φέρε και την εμπειρία του στον τομέα των μεταφορών. Υπάρχουν, ε, υπάρχει λοιπόν μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη στην οποία θα... Και τα σχόλια για το ΕΝΤΣΟ, το Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι τα ένας διαχειριστής μεταφοράς να προτείνει ένα έργο ενέργειας. Για μένα θα ήταν δραματικό αυτό. Επομένως, κατά την άποψή μου, είναι ε, και κλεισμένο των θυρών τα έργα αυτά βρουν σε ένα πολύ καλά ρυθμισμένο χώρο και κάθε βήμα καλύζουμε από την πλευρά Κομισιόν ότι εξελογούμε τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στα πιο φιλόδοξα σενάρια, στο πλαίσιο του πιο φιλόδοξου σενάριου από επίπεδο είναι να χρησιμοποιηθούν τα πιο φιλόδοξα σενάρια στην αξιολόγηση των έργων. Σε σχέση με τον αριθμό διαφορετικό μεθόδιο υπολογισμού και είχαμε σήμερα 95, στην πρώτη λίστα θα είχαμε περίπου 200. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία συζήτηση. Προσπαθώ να διατηρήσω μια ισορροπία στην Επιτροπή μας και να προσθέσω ότι είναι πάντοτε καλύτερο να χρησιμοποιεί κανείς αέριο παρά άνθρακα ή πετρέλαιο. Και γι' αυτό και το πολύ σημαντικό λόγο ξεκινήσαμε με τους από εργοστάσια αερίου. Προσπαθώ λοιπόν να διατηρήσω την ισορροπία σε όλες τις συζητήσεις μας, γιατί το να ρωτάτε ένα τόσο θεμελιώδες ερώτημα, όταν δηλαδή θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους ε, της Συμφωνίας των Παρισίων, Από με πολύ αριό, είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει φυσικά να μετακινηθούμε προς την αποθήκευση ενέργειας, γιατί τη χρειαζόμαστε. Και χωρίς ε, καλά αποτελέσματα στην αποθήκευση, φυσικά και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, βέβαια έχουμε και λίγο κατανόηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, ήταν πολύ καλή η συζήτηση, κυρία μου. Σε ένα χρόνο έχουμε και τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω ποια πολιτική ομάδα προτιμάτε. Τι ε, τις έχετε όλες εδώ ενώπιόν σας. Βλέπετε. Να πάμε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι η ενημέρωση για τον φορέα των Ευρωπαϊκών ε, Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες. Ο κύριος Τοσενόφσκι ήρθε να μας ενημερώσει, αλλά πρώτα πρώτα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ντελκαστίγιο όσον αφορά το code, τον κώδικα των επικοινωνίων. Σας ευχαριστώ, Φρεδρίας. Τώρα πάμε για την 1η Φεβρουαρίου. Ε, με την Βουλγαρική Προεδρία, πρώτη φάση. Όλο αυτόν τον καιρό προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάτι λόγο. Να δούμε τώρα μήπως 1η Φεβρουαρίου επί Βουλγαρικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε και να συμφωνήσουμε για κάποια επίμεχα ζητήματα. Και ίσως μπορέσουμε να κλείσουμε το κομμάτι του ζητήματος κατά τον δεύτερο τεμερή διάλογο της Βουλευτικής Προεδρίας το θέμα των η πρόσβαση στα δίκτυα. Άρα το θεματολόγιο παραμένει ζωντανό και θα πάμε μήπως κλείσουμε τέλη Απριλίου. Όλες οι πολιτικές ομάδες υποστήριζουν, επομένως έχουμε θέση αποφασιστική. του φάσματος. Οπότε να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες ε, για τη βοηθειά σε αυτή τη διαδρομική. Να ευχαριστήσω και την γραμματεία μας. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα, Εύγεν, για τον κανονισμό Μπέρεκ. Ευχαριστώ. Είναι στενή η σχέση ε, του Μπέρεκ, του κανονισμού Μπέρεκ τέλο πάντων, με αυτό το οποίο μας είπε η Πίλαρ Επομένω, ε, υπάρχει εδώ κοινή πορεία, κοινό χρονοδιάγραμμα και γι' αυτό και παρακολουθούμε τους τρεις διαλόγους που γίνονται για το code. Το Συμβούλιο έχει στάση που προσεγγίζει στην ε, δική μας και συμφωνούμε ότι χρειάζεται διτή, διπλή δομή στον κανονισμό Μπέρεκ ή τέλος πάντων στο, στο, στο φορέα αυτόν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε από πλευρά τη να συνεχίζουν να ισχύουν όσα ισχύουν σήμερα. Αλλά στο Κοινοβούλιο οι περισσότερε πολιτικέ ομάδε συμφώνησαν μαζί μα και ακριβώ με αυτά που είπαμε και στην Επιτροπή μα. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή προσέγγιση. Να δούμε αν θα ληφθούν αποφάσεις για το code που θα καλύψουν και το BEREC εάν τελικά υπάρξουν αλλαγές. Εκκρεμεί το θέμα των κατοξιδότηση παράξεων. που αφορούν το κόλτ και κατόπιν ε, ε, μεταβιβάστηκαν και στο Μπέρκ. Επίσης το θέμα είναι το ποιες θα είναι οι αρμοδίες αρχές και τα σχετικά. Εμείς Πάμε για πραγματεύση σε ακόμα έναν τριμερή διάλογο. Και ελπίζουμε τέλος Απριλίου θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδρομή και έτσι θα ευθυγραμμιστούμε και με τις εξελίξεις στο χρονοδιάγραμμα του Code. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όσο χρόνο το, το χρόνο που μας απομένει τέλος πάντων. Και πάλι ευχαριστήρια ε, προς την ε, πιλάρια της εργασίας της.